οι εκπρόσωπος που προσπαθούν συνεχώς να κάνουν κάτι από την κατάσταση που προέκυψε. Εάν προσπαθήσουμε λοιπόν μαζί έχουμε μια ευκαιρία. Εάν παριστάνουμε ότι κάνουμε κάτι βεβαίως δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Σας ευχαριστώ κύριε Φλέκενστάιν. Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Μπέλντερ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για μια ευρωπαϊκή τοποθέτηση απέναντι στην ε, περίπλοκη κατάσταση στη Λιβύη απαιτείται μια ευρωπαϊκή λεπτέστητη διπλωματία. Υπάρχουν εδώ πέρα διαφορετικά συμφέροντα, τουλάχιστον δύο διαφορετικές κυβερνήσεις και πάρα πολλές αμέτρητες ένοπλες ομάδες και Βλέπουμε πως ε, και εντός της ε, Ιταλικής ε, κυβέρνησης, έφυγε ο κύριος Καστάλντε, ότι υπάρχει διχασμός. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος κίνδυνος εδώ πέρα στη Λιβύη είναι οι τζιχαντιστικές ομάδες που σχετίζονται και με την Τουρκία. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πολιτική ε, περιορισμού της ε, κατάστασης και της κρίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπέλντερ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Κλοντ Μωρές. Κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Γιάλα Σέντερ και ο κύριος Καστάλτο και άλλοι σωστά περιέγραψαν την κατάσταση, τις παρεμβάσεις που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση η Αντιπρόεδρος είναι εδώ για να μιλήσει με αντιμετώπιση της ε, άμεσης ε, καταστάσεως και Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δηλαδή στην Επιτροπή μας πρόσφατα και αναφέρθηκε στις στρατηγικές που θέλει να εφαρμόσει. Τη ρωτώ, όπως και η κυρία Σπινέλη, πώς θα κινηθούμε με την επέκταση της ε, επιχειρήσεως Σοφία χωρίς να έχουμε σκάφια αρκετά υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας. Θα αλλάξουμε απόψεις αν επιδεινωθεί η κατάσταση. Είδαμε τα Ρίκα Σίλκα, πήγαμε στο στατόπεδο εκεί, όπως είπε η άλλα Σέντερ, είδαμε εκεί τους ε, διάφορους πρόσφυγες που είναι παγιδευμένοι. Ξέρουμε ότι αντιμετωπίζεται, είναι θέμα συνεργασίας. Έχουμε τον κίνδυνο χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες να έχουν παγιδευτεί σε κέντρα κράτησης, στο Κάζα Μπενκαζίρ, στο κέντρο κράτηση εκεί. Οι πληροφορίε που λαμβάνουμε και έχουμε επισκεφτεί και τη Λιβύη, όλα δείχνουν ότι είναι μια κρίση που θα μεγεθυνθεί λόγω αυτής της έντονης περίοδου. Ρωτάω ξανά, υπάρχει ευελιξία στον αφορά την προσέγγιση. Και πείτε μας, ποια είναι η κατάσταση αφορά την επιχείρηση Σοφία. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα, ο κύριος Γιούρεκ έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωπε, κυρίες και κύριοι. Ε, με την τραγωδία της Λιβύης έχουμε άλλη μια σκηνή αυτής της μεγάλης τραγωδίας που γίνεται στην άμεση γειτονία μας μαζί με την Αραβική Άνοιξη. Ε, σημαντικό και τραγικό πάθημα και δίδαγμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά κοινή ευθύνη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σχέση μας ε, απέναντι σε εταίρους εκτός της Ευρώπης ε, θα πρέπει να γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και συγκρίνοντας την πολιτική με θέματα στα οποία μπορούμε να προ... προτείνουμε κάποιες εναλλακτικέ λύσεις, αλλά όχι με βάση την ιδεολογία και τους ευσεβείς μας πόθους. Είδαμε την τραγωδία στη Συρία. Τώρα γινόμαστε μάρτυρες μιας αντίστοιχης τραγωδίας και κλιμάκωσης ε, στη Λιβύη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το συμφέρον του λιβικού λαού και να, ε, λάβουμε, να υπομισθούμε τις ευθύνες για, το, για τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιούρο. Η κυρία Κέγγι έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είναι ώρα τώρα για διχασμό και διαρέσεις. Η κόλαση της Λιβύης απαιτεί από όλου να υπομισθούμε τις ευθύνες μας. Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διεθνείς οργανισμοί, κυβερνήσεις εθνικές Υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αλλά θα πρέπει επίσης όλοι να συμβάλλουμε στην εξέβρεση πολιτικής λύσεως διαρκείας. Μια λύση που θα έχει σαν προοπτική μακροπρόθεσμη την ειρήνευση, τη σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση της χώρας. Ο απολογισμό όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή είναι πάρα πολύ βαρύ. Σαν στόχο έχουν τεθεί νοσοκομεία, σχολεία, ε, στατόπεδα προσφύγων ακόμα ευάλωτοι άνθρωποι. Πολλοί από αυτού είναι φυλακισμένοι σε μια κατάσταση με πολύ μεγάλο κίνδυνο και προσθέτονται εκεί αριθμός γυναικών, ανθρώπων και παιδιών, ε, ε, ανδρών και παιδιών που δεν μπορούν να τους αφήσουμε χωρίς προστασία διεθνή. Και την Ευρώπη κάποιοι τη θεωρούν σαν μια χώρα αποβίβασης ασφαλή και είναι αυτοί που κερδοσκοπούν με τι ζωέ των ανθρώπων για εύκολε εκλογικέ συμφωνίε. Τώρα περισσότερο πολύ οι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι υπεύθυνε και θα πρέπει να επιστρέψουμε στην επιχείρηση Σοφία. Ζητώ από την ύπατη εκπρόσωπο την ερώτηση αυτή. Θεωρείται ασφαλή χώρα η Λιβύη. Χρειαζόμαστε απάντηση. Και ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, Άλφρετ Σαντ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πέρα βλέπουμε πως πρέπει να επικρατήσει το συμφέρον του λαού της ε, Λιβύης. Πρέπει πρώτα απ' όλα λοιπόν να συμφωνήσουμε στα βασικά. Το βασικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μην είναι η Λιβύη μια αιστεία τρομοκρατίας. και κάποια στιγμή αργότερα αν υπάρξει σταθερότητα μπορεί να υπάρξει και δημοκρατία και ειρήνη. εντάξει. Δεν πρέπει να ανατρέπουμε καθόλου που δεν μας αρέσουν για το χύψη λόγο γιατί βλέπουμε ότι στην περίπτωση της ε, Λιβύης ε, το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο πρέπει λοιπόν καλή την πίστη να επιτρέψουμε σε όλες τις δυνάμεις ε, στην ε, Λιβύη να εκπροσωπηθούν. Και δεν μπορούμε βεβαίως να συνεχίσουμε να δεχόμαστε την παράλυση που υπάρχει ε, στην Λιβύη. Πρέπει να στηρίξουμε αυτούς που θέλουν να ενώσουν την χώρα για να σταματήσει η αναρχία, να υπάρξει ασφάλεια για τον λαό της Λιβύης και σταθερότητα. Αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει και η κοινωνία στη χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σαντ, κάτι πήρε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ε, και περισσότεροι ακόμα τραυματίστηκαν. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των τελευταίων μαχών ε, στην Λιβύη και όλα αυτά ενώ υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε προς μια κατεύθυνση ομαλοποίησης και ακόμα και εκλογών. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση στην Τρίπολη και τον στρατηγό ο δεν την υπακούει. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να ανεχτούμε αυτήν την κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική η οποία θα μας οδηγήσει στην εδραίωση τη διαδικασία της ε, Ειρηνή Αλλιώ. Ε, βλέπουμε ότι επικρατεί αναρχία και η χώρα γίνεται ένα πεδίο δράσης ε, τρομοκρατικών οργανώσεων. Πρέπει λοιπόν να αποσυρθούν τα στρατεύματα του στρατηγού, να υπάρξει η δυνατότητα να λειτουργήσουν οι συνομιλίε στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Μόνο έτσι θα ειρήνη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε κυρία Πύρη. Και... Περνάμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Παρακαλώ ένα λεπτό ο καθένας, γιατί έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας μέχρι το βράδυ. Ο κύριος Φαρία είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπατή, εκπρόσωπη, εκπρόσωπε. Η στρατική κλιμάκωση στη Λιβύη, πέραν των κοινωνικών συγκρούσεων που έχουμε και στη χώρα αυτή και στι γειτονικέ χώρε, έχει σοβαρέ οικονομικέ, ε, ανθρωπιστικέ συνέπειε και συνέπειε στην ασφάλεια. Γιατί έχουμε ένα νέο μεταναστευτικό κύμα. Ε, ε και τα επιχειρήματα αυτών που θεωρούν τη Λιβύη ασφαλή χώρα και χώρα μπορεί να δεχτεί επιστροφή. Και μάλιστα η ανθρωπιστική βοήθεια μερικών εκατομμυρίων ευρώ δεν θα πρέπει να μας εμποδίσει στο να λάβουμε μια κοινή θέση και να ζητήσουμε ε, άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών ε, και εκεχηρία στην πόλη και επιστροφή σε μια πολιτική συζήτηση μεταξύ του τον Μπρουκ και της Τρίπολης για να εξασφαλίσουμε ειρήνη και σταθερότητα για όλο το λιβικό λαό. Θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους ίδιους τους Λιβίους να ε, αναλάβουν την ευθύνη για το μέλλον τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φαρία. Η Άννα Γκόμες είναι η επόμενη ομιλήτρια. Αλλά δεν την βλέπω στην αίθουσα. Οπότε προχωράμε. Πατρίσια Λοράντο. Έχετε το λόγο. Merci. Ευχαριστώ. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, η κατάσταση στη Λιβύη είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Τουλάχιστον 150 άτομα έχασαν τη ζωή τους. 614 ε, τραυματίστηκαν και 18.000 εκτοπίστηκαν μετά την επίθεση του στρατηγού Χαφτάρ. Ε, έχουμε κατάσταση φιλίου πολέμου μετά την ανατροπή του Καντάφη το 2011. Και σίγουρα ο διχασμός μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπόδισε την ανέβρεση λύσης ε, στη σύραξη της Λιβύης. Και μάλιστα μερικές από τις ε, χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία είναι άμεσα υπεύθυνε για την κατάσταση. υπάρχει τεράστια απειλή για την ασφάλεια και την τάξη και οι τρομοκρατικέ ομάδε και οργανώσει στη Λιβύη εξακολουθούν να υπάρχουν. Και αυτό ο νέο εμφύλιο πόλεμο είναι μάνα εξ ουρανού για τι παραστρατιωτικέ ε, και ισλαμιστικέ δυνάμει. Κάτι που ίσω ε, μα οδηγεί σε ένα νέο κείμενο ε, μεταναστευτικών ροών και αποσταθεροποίηση και τη Τινησία που είναι πολύ κοντά. Ε, θα πρέπει να διευκολύνουμε μια επαναφορά στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων για την ανέβρεση ειρηνευτική λύση ε, με βάση την πραγματικότητα που επικρατεί στη Λιβύη για να αποφύγουμε ένα νέο αίματο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαλάντ. Και τώρα, Bill Etheridge. Ευχαριστώ. Η Λιβύη και όλη η κατάσταση αφορά την Αραβική Άνοιξη είναι ένα μάθημα για τη δυτική παρέμβαση σε χώρες που δεν κατανοούμε. Για μέρη που περισσότερο βλάβες προξενούμε, παρακαλώ. Κοιτάξτε, χάος έχει προκληθεί, πρόσφυγες, θάνατοι. Ποιος κερδίζει από όλα αυτά. Αν αυξάνονται οι δεσπότες, τρομοκρατικές ε, ομάδες ενισχύονται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στο μέλλον το να παρεμβαίνουμε μέσω μοβαρδισμών και στατιωτικών επεμβάσεων σε αυτά τα μέρη δεν θα είναι η λύση θα χειροτερέψει η κατάσταση. Πρέπει να είμαστε εκεί να μιλάμε με τον κόσμο, να βοηθάμε, να πραγματοποιούμε διπλωματικές επαφές, να εμπορευόμαστε. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι οι μέρες του μειωδών παρεμβάσεων νεοφιλελευθέρων πρέπει να μείνει στο παρελθόν. Μόνο το εμπόριο και οι συνομιλίες ανήκουν στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Έθριτς. Γέρι Πόσπισιλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά την ε, είπατε εκπρόσωπο και συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό πως μόνο πολιτική λύση μπορεί να υπάρξει. Η χώρα αποσταθεροποιείται και δυστυχώ δεν έχουμε μια πραγματική στρατηγική. κανεί ε, δεν ξέρει ποια συγκεκριμένα βήματα θα ήταν τα σωστά. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες διπλωματικές προσπάθειες και ελπίζουμε να αποδώσει η διπλωματία. Κυρία Μογκερίνη, η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη και φοβάμαι ότι εμείς μόνο μιλάμε εδώ πέρα και δεν κάνουμε τίποτα για να επιλύσουμε την κρίση. Γιατί η περαιτέρω ψωθεροποίηση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ περισσότερους πρόσφυγες που θα έρθουν στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Σας ευχαριστώ και πώς πες Κύριε Στρογεύσκη. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την εκτίμηση μου ε, για τις ενέργειες της ΥΠΑ της εκπροσώπου αλλά και το ειδικό επεσταλμένο του ΟΗΕ. Πιστεύω ότι ο πολιτισμένος κόσμος θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί και κάνει ό,τι μπορεί για την κατάσταση. Αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι την γνώση, την καλύτερη και πιο συγκεκριμένη γνώση. Η έλλειψη πληροφοριών ε, μας οδηγεί σε έκπληξη, σε φινιδιασμό, σε απογοήτευση. Μερικές φορές υφιστάμεθα και οικονομικές σημείες. Ε, μερικές φορές νιώθουμε τελείως ανήμποροι απέναντι στην κατάσταση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα των πληροφοριών για να έχουμε καλύτερη γνώση και ε, στο μέλλον να είμαστε πιο συνεπείς και πιο αποτελεσματικοί. Επανειλημμένος ε, έλαβα το λόγο για πολλά θέματα εξωτερικής πολιτικής, για τις συγκρούσεις στην Αφρική, για τις συγκρούσεις στην Αγγής Ανατολή. Όλα αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Το γεγονό δηλαδή ότι εκφράζουμε την έκπληξή μα, τον ευνηδιασμό μα, τη δυσάρεστη έκπληξη για αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Όχι. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη ενημέρωση, θα πρέπει να βελτιώσουμε τι γνώσει μα για την κατάσταση για να μην ευνηδιαζόμαστε. Έχουμε δυσάρεστε εκπλήξει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Στρογεύσκη. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών στο ΚΑΤΣΔΙ. Θα ξαναδώσω το λόγο στην ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τη λύπη μου που συνάδελφοι, που, κάποιοι ευρωβουλευτές που έθεσαν ερωτήσεις εγκατέλειψαν την αίθουσα και δεν θα ακούσουν τις απαντήσεις. Ε, όταν συζητούμε ένα τόσο σοβαρό θέμα, δεν εκφράζουμε καμία έκπληξη ευνηδιασμό. Χρόνια ολόκληρα συζητάμε αυτό το θέμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη και το συζητούμε με εταίρα μας στην περιοχή, με τον Αραβικό Σύνδεσμο, με την Αφρικανική Ένωση. Αυτό που με είναι σε αυτήν την τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τις ευρωεκλογέ ότι έχουμε περισσότερους ε, θεατές στους εξώστες των επισκεπτών παρά ευρωβουλευτές στην αίθουσα της Ολομέλειας για τη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ε, έπαινος για όλους όσοι είστε παρόντες τελικά στη συζήτηση. Και ευχαριστώ για την υποστήριξη του έργου μας τις τελευταίες εβδομάδες που δεν ήταν καθόλου εύκολο και το, τις προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή θέση για τα θέματα αυτά, κάτι που δεν ήταν εύκολο να έχουμε σύγκληση. Σήμερα όμως έχουμε μια ενωμένη ευρωπαϊκή πολιτική και δράση. Θέλουμε να σταθεροποιήσουμε τη χώρα δίνοντας την ευκαιρία στον ίδιο τον Λιβυκό λαό, στους ίδιους τους πολίτες της Λιβύης, ε, στους ενδιαφερόμενους, στους συμβαλόμενους, στους διάφορους φορείς και οργανώσεις, όσο ευάλωτοι και αν είναι, όσο συγκρουσιακοί και αν είναι μερικές φορές, ε, δίνουμε την ευκαιρία στους λιβικούς φορείς να βρουν το δικό τους δρόμο προς μια ενωμένη χώρα για την ενωμένη τους πατρίδα. Και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που παρήχε στις προσπάθειές μας και πιστεύω ότι χάρη στη συνεργασία μας έχουμε καταφέρει και στις δύσκολες αυτές συνθήκες μερικά θετικά πράγματα. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για δύο τινά. Καταρχήν για την υποστήριξη που μονίμως προσφέρουμε στα Ηνωμένα Έθνη και στους δικούς απεσταλμένους των Ηνωμένων Εθνών και μπορούν να υπολογίζουν στην αμέριστη υποστήριξή μας την πολιτική, οικονομική, διπλωματική, την υποστήριξη επιτόπου και νιώθω υπερήφανη για το γεγονό ότι οι δικοί μα υπάλληλοι πήγαν στην Τρίπολη και επέστρεψαν στην Τρίπολη πολύ νωρίτερα από το προσωπικό άλλων διεθνών οργανώσεων. Ε, βέβαια η κατάσταση έχει αλλάξει πρόσφατα. Θα επιστρέψουν πάντως, ελπίζω να επιστρέψουν ε, ως ο Νούπο στην Τρίπολη και να έχουμε και νέα εγγένεια το γραφείο μας στην Τρίπολη μετά από μακρά απουσία μας από την πρωτεύουσα. Και περιμένουμε με αγωνία αυτή την ε, αποκατάσταση της ομαλότητας στο μέτρο του δυνατού, γιατί η απόλυτη ομαλότητα στη Λιβύη τέτοιου χαλεπού καιρού δεν την προβλέπω, αλλά τουλάχιστον κάποια ομαλότητα. Πάντω είναι σημαντικό και ο Λιβυκό Συνάδελφο να γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά τη όργανα ανέκαθεν προσπαθούσαν να βοηθήσουν με επικοδομητικό και έντιμο τρόπο και οικονομικά, αλλά και πολιτικά και διπλωματικά. Και αυτό συνέβη χάρη και στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το δεύτερο πράγμα για το οποίο νιώθω υπερήφανη σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον είναι το έργο που καταφέραμε επιτέλους να ξεκινήσουμε και θα πρέπει να παγιώσουμε στο μέλλον, να το εδραιώσουμε περαιτέρω για τα κέντρα κράτησης, να τα κενώσουμε και να τα κλείσουμε σε συνεργασία με τις οργανώσεις ε, ε, των Ηνωμένων Εθνών. Και παραλαμβάνω, η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με τους Λιβύους μαζί και όχι ερήμην της Λιβύης. Γιατί αν έχουμε κλιμάκωση της ένοπλης σύραξης στη Λιβύη, το πρώτο μου μέλημα είναι οι ανθρώπινες ζωές που θα χαθούν και η επιδείνωση της προοπτικής του πολιτικού διαλόγου. Δεν με φοβίζει τόσο ο κίνδυνος ο μεταναστευτικός προς την Ευρώπη. Ο, προβληματίζει ο κίνδυνος για τη ζωή των ίδιων των μεταναστών. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους που το τόνισα, γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε ως μέλημά μας τη ζωή ε, των μεταναστών, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, η ανθρώπινη ζωή πρώτα απ' όλα. Και μετά να βοηθήσουμε τη Λιβύη και το λιβικό λαό. Γιατί η Λιβύη είναι μια ε, χώρα εταίρος και μια γειτονική χώρα και θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως τέτοια, ως εταίρο και ως γειτονική χώρα. Και πρόσφατα έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με τα, τον ΟΗΕ, με την Υπατήρμοσία για τους πρόσφυγες, με την Αφρικανική Ένωση για να αντιμετωπίσουμε το, τη λαθροδιακίνηση ανθρώπων και την εμπορία ανθρώπων και βοηθήσαμε τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και καταφέραμε να κενώσουμε 40.000 ε, τέτοιους μετανάστες και πρόσφυγες από τα κέντρα κράτησης, είτε ε, ε, προς τα κέντρα της ΥΠΑ της Αρμοστίας που ε, είναι καλύτερα προστατευμένοι είτε να τους ε, επαναπατρίσουμε στις χώρες προέλευσής τους με τη συνεργασία και της Αφρικανικής Ένωσης και των κρατών μελών της. Όλο αυτό το έργο, όπως σας είπα, έγινε σε μια κατάσταση με μια στρατιωτική κλιμάκωση και μια αυξανόμενη ανασφάλεια που καθιστά τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Και Συμφωνώ με την έκκληση που απέθυνε ο Φιλίππο Γκράντιο, το αρμοστής για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών, να εξασφαλίσουμε πρόσβαση ε, στο προσωπικό του, της ΥΠΑ της Αρμοστίας προς τα κέντρα κράτησης, να ανοίξουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ζωτική σημασία για να διασφαλίσουμε τη ζωή των προσφύγων και μεταναστών στα κέντρα αυτά. Μερικοί ε, με ρώτησαν ε, κάτι που αφορά περισσότερο το γενικότερο μας έργο για τη μετανάστευση παρά τη Λιβύη. Δεν θεωρούμε τη Λιβύη ασφαλή χώρα σε καμία περίπτωση. Αυτό το έχω πει και εγώ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επανειλημμένω μάλιστα. Και η κατάσταση, η κρίση αυτή δεν έχει αλλάξει και είναι προφανέ μάλιστα με τι παρούσε συνθήκε ότι η Λιβύη δεν είναι ασφαλή χώρα. Κάποιοι ευρωβουλευτέ με ρώτησαν για την επιχείρηση Σοφία. Ε, όπως ξέρετε και δεν είναι κανένα μυστικό, εγώ πρότεινα στα κράτη-μέλη όχι να αποσύρουν τα πλοία τους. Εγώ είπα να παραμείνουν τα πλοία στα διεθνή χωρικά ύδατα, γιατί ήταν πολύ σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας για τους λαθροδιακινητές. Και αν ε, οι αφήξει από τη Λιβύη στην Ιταλία μειώθηκαν πάνω από 80% την τελευταία διετία. Αυτό έγινε χάρη στην παρουσία των πλοίων ε, στα πλαίσια της επιχείρησης Σοφία στη θάλασσα. Και φυσικά βλέπουμε την αντίφαση το να έχουμε μια ε, ναυτιλιακή επιχείρηση χωρίς να έχουμε πλοία. Βέβαια, ε, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν κάτι διαφορετικό τελικά. Ελπίζω να αναθεωρήσουν την απόφασή τους και τελικά να μεταπιστούν και να ξαναφέρουν τα πλοία τους στα διεθνή χωρικά ύδατα. Γιατί υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες έχει νόημα αυτή η παρουσία των πλοίων. Όχι μόνο για να αποτρέψουμε τους λαθροδιακινητές και τους εμπόρους ανθρώπων, αλλά ε, και για να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και τα καθήκοντά μας και να εφαρμόσουμε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας σε ό,τι αφορά το εμπάργο πετρελαίου και όπλων και το σχετικό έλεγχο. Και πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί αν έχουμε αυτιλιακή παρουσία στη θάλασσα, στα διεθνή χωρικά ύδατα. Και επαναλαμβάνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω και δημοσίως, το έχω ήδη πει και ανοιχτά και δημοσίως. Πιστεύω ότι χωρίς ε, πλοία, χωρίς ναυτιλιακή παρουσία, η επιχείρηση Σοφία δεν πρόκειται να υλοποιήσει αποτελεσματικά και πλήρω την εντολή τη. Και ελπίζω τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν την απόφασή του να αποσύρουν τα πλοία του. Και νομίζω ότι είναι ευθύνη και επιλογή του και ελπίζω να μεταπιστούν τελικά και να αναθεωρήσουν την απόφασή του στο εγγύ μέλλον. Θα ήθελα εν κατακλείδη να πω ότι ευχαριστώ και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλες τις πολιτικές παρατάξεις για την υποστήριξή τους στο έργο της ΕΙΕΔ και την ε, έκκληση που απέφθαιναν τα τελευταία μήνες ε, και τη συμπαράσταση προς τις προσπάθειες και του ΟΗΕ. Θα πρέπει να, να επιστρέψουμε σε μια πολιτική διαδικασία στην οποία ε, θα πρωτοστατεί η ίδια η Λιβύη, ο Λιβικός λαός και τα ενδιαφερόμενα μέρη και να αποκλιμακώσουμε αυτές τις στρατιωτικές εντάσεις που δημιουργήθηκαν, να καταπαύσουμε να έχουμε κατάπαυση των εχθροπραξιών και να δημιουργηθούν ισχυροί ειρηνικοί θεσμοί στη χώρα. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι παρά τις λίγες φωνές που ζήτησαν κάτι αντίθετο, οι περισσότεροι ζήτησαν ανοιχτούς ανθρωπιστικούς διαδρόμους για παροχή κατεπίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, άμεση κατάπαυση του πυρός και των εχθροπραξιών και επαναφορά στην πολιτική συζήτηση και στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της Διεθνούς Συνδιάσκεψης υπό την αιγύδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να διαφυλάξουμε την ελπίδα του λιβικού λαού ε, να έχουν μια ειρηνική και ομαλή χώρα και ένα ε, μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Υπάτη εκπρόσωπε. Και τώρα θα πάρει το λόγο η εκπρόσωπος ε, της Ένωσης για το θέμα της ε, ε, αναγνώριση από τη ΣΥΠΑ των υψηπέδων του Γκολάνου στου ελληνικού εδάφους και πιθανή προσάρτηση των οικισμών τη Δυτική Όχθη. Κύριε Μογκερίνη, είναι δύο χωριστά θέματα. Και τα δύο είναι επίπτωση του πολέμου του 67, αλλά είναι χωριστά. Από τη μία πλευρά έχουμε την απόφαση τη ε, κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναγνωρίσει τα υψώματα του Γκολάν ω ε, Ισραηλινού εδάφου και η άλλη είναι η πολιτικισμών τη ελληνική κυβέρνηση στη δυτική όχθη. Θα αντιμετωπίσω λοιπόν τα δύο θέματα χωριστά. Πρώτον, η αναγνώριση του υψηπέδων του Γκολάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σαφή και σαφή θέση, την οποία είχα την ευκαιρία να επαναλάβω σαφέστατα επανειλημμένα και πρόσφατα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει η Ισραηλινή κυριαρχία επί εδαφών τα οποία κατέχει από τον Ιούνιο του 1967 με βάση το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα 2.42 και, ε, και 2.79 και αυτό αφορά και τα υψήματα του Γκολάν. Το Μάρτιο έκανε μια δήλωση από πλευρά των 28 κρατών μελών, διευκρινίζοντα ότι αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καθεστώς των ψηφίσματος του Γκολάν. Αυτή ήταν πάντα η θέση μας και δεν έχει αλλάξει. Παράλληλα, τα πέντε κράτη-μέλη της Ένωσης που είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία εξέφρασαν την κοινή του θέση αυτή σε μια κοινή δήλωση που έκαναν στη Νέα Υόρκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, όντω λοιπόν για το θέμα αυτό, μιλούν μια φωνή όπω πάντα ζητάμε. Και δεν είναι το μόνο θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω τα πέντε κράτη-μέλη λοιπόν, που είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας αυτή τη στιγμή, γιατί η πρακτική αυτή συντονισμού θέσεων και κοινή έκφραση των θέσεων αυτών και με δημόσιε δηλώσει προ τον τύπο από τα πέντε κράτη και επίσης σε συναντήσει και με μένα για να συντονίσουμε τη θέση των κρατών μελών στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτή η πρακτική γίνεται όλο και πιο συχνή και αυτό νομίζω είναι και ευθύνη μας να στηρίξουμε το πολυμερές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες. Σε αυτή τη συγκυρία. Τώρα, το δεύτερο θέμα είναι η πολιτική επικισμού της Ισραηλινής κυβέρνησης δεν θα σχολιάσω τι ε, πρακτικέ ε, μπορεί να ακολουθήσει τώρα η κυβέρνηση που επροέκυψε μετά τι εκλογέ, που ακόμη δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί, αλλά αυτό που διαπιστώνουμε πρόσφατα, δηλαδή του τελευταίου μήνε, είναι ότι οικοδομούνται και περαιτέρω επικισμοί. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύθηκαν ε, σχέδια για 4.000 επιπλέον κατοικίε αμέσω μετά. Κάναμε μια δήλωση όπου αναλάβαμε ότι όλοι οι επικισμοί είναι παράνομοι με βάση το διεθνέ δίκαιο και οι επικισμοί αυτοί μειώνουν τη βιωσιμότητα μιας ε, λύσης ε, δύο κρατών. Όχι μόνο απομακρύνεται αυτή η λύση, στην ουσία κομμάτι-κομμάτι αποσυναρμολογείται. Είναι λοιπόν σημαντικό ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει σαφώς ότι η εγκατάλειψη της λύσης δύο κρατών θα αυξήσει το χάος, όχι μόνο στους Αγίους Τόπους, αλλά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή που ήδη αντιμετωπίζει μεγάλες δυσχέρειες γιατί έχουμε πολλέ κρίσει ε, στην περιοχή που εξαπλώνονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Η επόμενη κλιμάκωση τη βία στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη πολύ εύκολα μπορεί να ξεφύγει από, να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και να έχει τραγικέ επιπτώσει σε μια περιοχή τόσο ασταθή όπω είναι σε αυτή τη φάση η Μέση Ανατολή. Επίση, η λύση με δύο κράτη και η δημιουργία ενό Παλαιστινιακού κράτου κατά συνέπεια για την κοινή γνώμη του αραβικού κόσμου θα είχε πολύ θετική επίπτωση σε μια περιοχή, παραλαμβάνω, που έχει αντιμετωπίσει τρομερέ ε, αναταράξει τα τελευταία χρόνια. Πρέπει λοιπόν η προοπτική δημιουργία δύο κρατών να παραμείνει ζωντανή και να διατηρήσουμε τη δυνατότητα να υπάρξουν νέε διαπραγματεύσει για την επίτευξη ειρήνη. Ούτω ώστε να είμαστε ρεαλιστέ και επιτυχεί οποιοδήποτε σχεδιασμό για το μέλλον των σχέσεων Ισραήλ και Παλαιστίνη θα πρέπει να ξεκινήσει με βάση τις ε, διεθνείς αναγνωρισμένα αναγνωρισμένες παραμέτρου, δηλαδή τα όρια του 67 με αμοιβέ αλλαγέ, εδαφών και η Ιερουσαλήμ να είναι αναγνωρισμένη πρωτεύουσα των δύο κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιμείνει σε αυτή τη θέση και θα συνεχίσει να το επιμένει. Θα αναγνωρίσουμε αλλαγές των συνόρων του 1967 πριν δηλαδή από την σύγκρουση, αν υπάρξει συμφωνία των δύο μερών σε σχέση με την Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η θέση αρχή. Αλλά βασίζεται και σε μια ρεαλιστική εκτίμηση τη κατάσταση επιτόπου. Διότι η λύση των δύο κρατών είναι πρώτα απ' όλα ουσιώδη για την επίτευξη ειρήνη, αλλά και για την ασφάλεια. Την ασφάλεια του Ισραήλ πρώτα απ' όλα. Είναι ουσιώδη για τη δημοκρατία και στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Είναι απαραίτητη για να υπάρξει πραγματικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίου. Και να προσθέσω, ακόμη πιο σημαντικό, είναι αναγκαία για την ειρήνη, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρη τη περιοχή, άρα και των γειτονικών χωρών. Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, θα επιδεινωθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα όπω την είδαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και σε αυτού του ε, χαλεπού καιρού. Νομίζω ότι η διατήρηση αυτή τη προοπτική είναι η πιο θαραλέα και η πιο επικοδομητική συμβολή που θα μπορούσαμε να έχουμε και η καλύτερη υπηρεσία προς την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει τους επόμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργαζόμενοι με όσους είναι διατεθειμένοι να εργαστούν για μια διαρκή, δίκαια και βιώσιμη ειρήνη. Πρώτα απ' όλα με τους ε, Άραβες εταίρους μας, τους τελευταίους μήνες, είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με την ηγεσία του Αραβικού Συνδέσμου, των χωρών του Αραβικού Συνδέσμου, στην πρώτη συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αραβικού Συνδέσμου στην Αίγυπτο και με τη δική μου συμμετοχή στη δεύτερη, συγγνώμη, στην τρίτη συνάντηση κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου. Και πρέπει να σας πω ότι η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λύση δύο κρατών αλλά και για τα υψίπεδα του Γκολάν ήταν από τα κύρια στοιχεία συζήτησης και είναι μάλλον από τα κύρια στοιχεία που βρίσκουν τους Ευρωπαίους και τους Άραβες ε, σύμφωνους σε αυτή την ε, δύσκολη συγκυρία. Οπότε θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, τόσο σημαντικό για την ασφάλεια και την ειρήνη στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, είπατε, είπατε εκπρόσωπε. Και τώρα θα παρακαλέσω εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να λάβει το λόγο ο κύριος Κριστιαν Πρέντα για ένα λεπτό. Είπα ότι εκπρόσωπε η ομάδα μου τάχθηκε κατά της διεξαγωγής της συζήτησης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει σαφή θέση σε σχέση με τα υψίπεδα του Γκολάν. Δεν αναγνωρίζουμε παρά μόνο αυτά που ορίζουν τα ψηφίσματα των ΕΕ 242 και 197 ε, σε σχέση με θέματα κυριαρχίας στα υψίπεδα του Γκολάνια. Μια απόφαση λοιπόν της κυβέρνησης Τραμπ δεν αλλάζει τίποτα ε, σε σχέση με την κατάσταση αυτή. Η δε δήλωση της 6ης Απριλίου η σχετική με την Δυτική Όχθη έγινε μόνο στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του Ισραήλ. Δεν υπήρχε ένας λόγος να υποστηριχθεί η προεκλογική εκστρατεία και ρητορική της άκρας αριστεράς εδώ στο Κοινοβούλιο, γιατί αυτό μόνο θα πλήξει την ε, εικόνα του Κοινοβουλίου αλλά και την διαδικασία για την ειρήνη. Αν πρέπει κάτι να πούμε θα πρέπει να είναι η διαπίστωση πως έχει καταρρεύσει το Συριακό κράτος και ότι υπάρχουν προβλήματα και σε σχέση με τα εψίπαδα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα και τις ιδιαίτερε ευαισθησίες που, ε, που έχει και το κράτος του Ισραήλ σε σχέση με τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στα ψήπαδα του Γκολάν με την υποστήριξη του Ιράν και κυρίως τη Χεσμολά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, κυρία Βαλενσιάνο, ένα μισή λεπτό. Είναι αλήθεια ότι αυτό που συμβαίνει ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη και τον δρόμο που ακολουθεί η κυβερνηση Τραμπ, Τράμπα, χέρι-χέρι με τον κύριο Γιονιτανιάχου, δεν είναι τίποτα το καινούριο. Είναι σαφές αυτό που κάνουν. Ακόμα και αν τον εκπλήσει τον κύριο Πρέντα. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. γιατί συνεχίζουμε να είμαστε πολύ δειλοί στην καταγγελία αυτού που είναι μια παράβαση της, του, του, διεθνούς δικαίου. Το ότι εμείς το ότι εμείς εκχωρούμε στην κυβέρνηση του Ισραήλ και της Αμερικής, στην κυβέρνηση της Αμερικής ε, είναι εκτός νόμου. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να του τιμωρούμε επειδή δεν τηρούν το διεθνές δίκαιο και άλλους να απευθύνουμε να μην το τηρούν. Ε, γιατί είμαστε τόσο δειλοί, γιατί έχουμε μια ε, κυβέρνηση αμερικανική που είναι σαφώς εχθρική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότερες παρεμβάσεις ε, που έχουν γίνει εδώ, οι περισσότερες ε, μου νομίζω παρεμβάσεις εδώ σε αυτή την ε, αίθουσα ήταν σε σχέση με το Παλαιστινιακό. Και αυτή είναι η τελευταία μου παρέμβαση. Πάλι μιλάμε για την αποτυχία της συνευτικής διαδικασίας. Είναι μια διαδικασία που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, που παράγει τεράστιες αδικίες και που δεν επιτρέπει τη λύση των δύο κρατών. Εμείς συνεχίζουμε από πολιτικής άποψη να το στηρίζουμε, αλλά από πρακτική απόψη δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό και θα πρέπει λίγο να υψώσουμε τη φωνή μας. Σας ευχαριστώ κυρία Βαλενσιάνο. Επόμενος ομιλητής εξ ονόματος της ομάδας της είναι ο κύριος Μπάς Μπέλντερ. Για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, Εάν έχετε επισκεφθεί το υψίπεδο του ΛΑΝ, γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το σημείο για την ασφάλεια του Ισραήλ και τους πολίτες της. Αν έχετε επισκεφθεί την περιοχή, θα ξέρετε ότι κοντά στη Συρία υπάρχει παρουσία ε, Χεσμολά και ε, το Ιράν μέσα στη στρατιωτική του δύναμη. Θα γνωρίζετε πως είναι τροποκράτες σύμμαχοι που θέλουν να εξαλείψουν από το χάρτη το εβραϊκό κράτος. Αυτό έχουν πει οι Ιρανοί. Έχουμε το αμερικανικό μοντέλο της αναγνώρισης του υψηπέδου του Γκολάν ως ε, ε, Ισραηλινό έδαφος και είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι με την Χεσμολά παρούσα εκεί θα πρέπει να ε, επικρατήσει ειρήνη με άλλους τρόπους. Εάν έχετε επισκεφθεί τα υψίπεδα του Γκολάν θα γνωρίζετε πόσο η, βιβλικές, πόσο η βιβλική σύνδεση υπάρχει του Ισραηλινού κράτους, του Εβραϊκού κράτους με αυτό το συγκεκριμένο μέρος. Θα πρέπει να πάψουμε να ερμηνεύουμε επληκτικά το διεθνές δίκαιο και να αναγνωρίσουμε τα υψίπεδα του Γκολάν ως εβραϊκά εδάφη όπως κάνουν και οι σύμμαχοι σύμμαχοι, κυρία Βαλενσιάνο. Αυτό κάνουν οι σύμμαχοι. Σας ευχαριστώ κύριε Μπέλτερ. Εκ μέρους ομάδας των Φιλελευθέρων η κυρία Βάουτμανς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είπατε εκπρόσωπε, αισθάνομαι βαθιά ανησυχία για την κατάσταση στο Ισραήλ. Είναι όλο και περισσότερα τα σημάδια που δείχνουν πως το Ισραήλ έχει εγκαταλείψει πλέον την ιδέα των δύο κρατών. Ο Νετανιάου θέλει να επεκτείνει το εδάφι της χώρας του, ε, επεκτείνοντας τους επικισμούς και τις προσαρτήσεις εδαφών. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή όπου η ειρηνευτική διαδικασία έχει εγκαταλειφθεί ουσιαστικά. Οι Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής είχαν στο παρελθόν συμμετοχή στην οικοδόμηση της ειρήνης. Ωστόσο σήμερα έχουμε την εντύπωση πως όλο και περισσότερο αποσκοπούν στην ε, αποδοχή παραβιάσεων του διεθνούς ε, δικαίου εάν δεν το παραβιάζουν οι ίδιοι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Γι' αυτό λοιπόν είπατε εκπρόσωπε θα ήθελα να σας ζητήσω να προβείτε σε ακόμη πιο σαφή διαβήματα σε σχέση με, την, ε, με τις δικές μας θέσεις. Είμαστε υπέρ όπως πάντα τις θέσεις δύο, για τη δημιουργία δύο κρατών ε, με βάση τα, τη διαχωριστική γραμμή τα σύνορα του 1967 κατά τρόπο βιώσιμο και περιμένουμε να αλλάξει η θέση του Τραμπ να μας πει τι είδου σχέδια αναπτύσσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ξέρω ότι σας έχουν αποσταλεί επιστολές από τις κυβερνήσεις των κρατών όλης της Ευρώπης. Θα θέλαμε να δούμε ακριβώς τι σας προτάθηκε και σας παρακαλώ να εκπροσωπήσετε από ακόμη πιο ξεκάθαρα την θέση αυτή, τη μόνη βιώσιμη λύση ε, των δύο κρατών. Και σας, σας παρακαλώ να διαβάσετε με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία ε, αναφέρουν αυτές οι επιστολές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βάουτμαντς και τώρα εκ μέρους της ΓΚΟΥ η κυρία Μαρία... Μαρίζα Ματίας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι τίποτα από αυτά δεν είναι καινούριο, αλλά όλο ένα και περισσότερο αφισβητείται η διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Είναι αλήθεια ότι η προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών ήδη υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή ε, ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ ε, δεν ε, ασχολείται καν. Εγώ συμμερίζομαι τη θέση μας, κυρία Μογκε... στη θέση σας, κυρία Μογκερίνη, αλλά έχουμε και άλλα μέσα. τι, θα, τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να έχουμε και άλλα μέσα στη διάθεσή μας. Υπάρχουν συμφωνίες σύνδεσης. Ας τις αναστείλουμε, ε, ας αποφασίσουμε αν θα τις αναστείλουμε ή όχι. Η υπεράσπιση των συνόρων του 67, συμφωνία ειρήνευσης, είναι μόνο λόγια σε ένα χαρτί ή πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά υπόψη να υπάρξει μια ε, συμφωνία και να κάνουμε, ασκήσουμε το κύρος μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρέντα, την ημέρα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρήθηκαν, θεωρούνται κάτι το, που, δεν είναι φυσιολογικό, τότε θα έχουμε πολύ ε, μεγάλο πρόβλημα. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να μας απασχολεί διαρκώς. Εγώ, μένα δουλειά μου είναι η περάσπιση αυτών των δικαιωμάτων. Κυρία Ματίας, εδώ δεν ερχόμαστε για να φωνοσκούμε αγαπητοί συνάδελφοι από την άλλη πλευρά της αίθουσας. Μπορείτε να στήσετε το λόγο με μία μπλε κάρτα, αν θέλετε κάτι να πείτε στην κυρία Ματία. Η κυρία Άουκεν, παρακαλώ, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σα και για τη σαφή γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Μέχρι τώρα όμω δεν κοστίζει τίποτε στο Ισραήλ το ότι συνεχίζει ε, μονομερή ε, κατάσταση κατοχής και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πλέον από τα λόγια να περάσουμε στις πράξεις για τις επιστολές που έγινε λόγος νωρίτερα. Οι Υπουργοί των Εξωτερικών και Πρωθυπουργοί των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν απερίφραστα ότι πλέον κάτι πρέπει να γίνει και ε, παραπέμποντας το ψήφισμα 2334 των Ηνωμένων Εθνών μιλούν για διαφοροποιημένη προσέγγιση ε, διαφορετική γλώσσα δηλαδή και αυτό σημαίνει ότι σταματούμε κάθε επικοινωνία με τους παράνομους επικισμούς, δεν πρόκειται για υπηρεσιακές επαφές και συναλλαγέ, δεν πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα κτλ. Να κλείσουν τελείω οι για του επικισμού. Ε, ένα τίμημα το οποίο με βεβαίω ότι αν έχει κάποιο κόστο για τους φίλους μας ε, στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη μπορούμε να του στηρίξουμε ώστε να μην χάσουν τίποτα και να μπορούν να προχωρήσουν μετά στην ειρήνη. Δεν βοηθούν τα λόγια πια και νομίζω το έχετε αντιληφθεί και εσεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άουκεν. Και τώρα παρακαλώ να συνεχίσουμε με τους ομιλητές μας των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Αγενά έχει τον λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είπατε εκπρόσωπε, η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Εξωτερική απέχει όσο ποτέ από αυτή από τις επιλογές της Αμερικανικής κυβέρνησης στην εξωτερική της πολιτική. Όταν εσείς υπερασπιστήκατε συμφωνίες με το Ιράν, είδαμε ότι κράτησαν αποστάσεις οι Πολιτείες. Με την COP21 είδαμε ότι κράτησαν αποστάσεις οι Πολιτείες. Τώρα με το Ισραήλ, βεβαίως οι Πολιτείες υποστηρίζουν τις πιο ακραίες τάσεις της κυβέρνησης του Ισραήλ ε, επιλέγοντας καταρχάς την ε, μετατόπιση της ε, πρεσβείας τους και αναγνωρίζοντας έτσι την, τα Ιεροσόλυμα ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Και τώρα έχουμε μια απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ για τα υψίπεδα του Γκολάν με την ευκαιρία της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες παραγνωρίζουν πλήρω το διεθνέ δίκαιο και τι αποφάσει των Ηνωμένων Εθνών. Και τώρα έχουμε μια απόφαση για εμπορικέ συναλλαγέ με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ένα κράτο ε, αλήτη που βλέπουμε να παραβιάζει κάθε έννοια ε, πολυμερούς ε, εμπορίου. Κυρία Είπατε ε, οι εκπρόσωπε, κάνατε ό,τι μπορούσατε, ό,τι έχετε σαν μέσα στα χέρια. Είτε πρόκειται για διπλωματία, είτε πρόκειται για αυστηρή γλώσσα. Αλλά υπάρχουν και δύο μέσα που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Συμφωνίε σύνδεση και εμπορικέ συναλλαγές Δύο τύπων κυρώσει δηλαδή, που μπορούν, ε, δύο τύπους κυρώσεων δηλαδή, που μπορούν ε, να αναγνωρίσουν τα κράτη αυτά έτσι ώστε να αντιληφθούν ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε ε, στις καλένδες τη λύση των δύο κρατών ώστε να εγκαταλείψουν και οι Ισραηλινοί αυτή την στάση σε σχέση με την κατοχή αλλά και οι Παλαιστίνοι την ορολογία της βίας και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει εμείς να σκόσουμε το λάβαρο της λύσης των δύο κρατών. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ. Ο, κύριο Πρέντα, ο κύριος Πρέντα, κυρία Αρένα, έχει ζητήσει μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Δέχεστε? Τι δέχεστε, ωραία. Παρακαλώ, κύριε Πρέντα. Μισό λεπτό, κύριε Πρέντα. Αγαπητή Μαρία, είπες ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι κράτος ανεξέλεγκτο. Δεν θεωρείς ότι τέτοιες τοποθετήσεις κάνουν ζημιά στις σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. δεν θεωρείς ότι και η αριστερά της ε, πολιτικής ομάδα και η ακροαριστερά είναι επίσης υπεύθυνε για την ε, επιδίνωση αυτής της ε, καλή συνεργασία και της σωστή ατμόσφαιρας στη σχέση με τις ΗΠΑ. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, μέχρι πού πρέπει να εκνευρίζουμε τους Αμερικανούς. Παρακαλώ απαντήστε. Αγαπητέ Ντάν, αγαπητέ κύριε Πρέδα, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν περίμεναν την Ευρωπαϊκή Αριστερά για να καταπατήσουν το διεθνέ δίκαιο. Όταν ο κύριο Τραμπ αποφασίζει να βάλει δασμού στο αλουμίνιο για να απαγορεύσει την εξαγωγή προ τι Ηνωμένε Πολιτείε αλουμινίου για λόγου ασφαλεία, αυτό σημαίνει ότι καταπατά το διεθνέ δίκαιο και τι διεθνεί συμφωνίε. Όταν αναγνωρίζουν ε, τα υψίπεδα του Γκολάν ω ε, Ισραηλινό έδαφο, παραβιάζουν ε, το διεθνέ δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά φταίει αυτή προκαλεί την κατανόηση μεταξύ ε, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Με συγχωρείς, αν εσύ θες να κάνεις ρεβερέντζες στον Τραμπ, αυτό δεν είναι πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η διαδικασία Catch the Eye έχουν υποβληθεί αρκετά αιτήματα. Θα πρότεινα την εξή λογική, γιατί Έχουμε πολλές ε, αιτήσει και έχουμε και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να πω ότι όσοι πήραν το λόγο στην ε, προηγούμενη ζήτηση Catch δεν θα πάρουν το λόγο τώρα. Και δεν θα δώσω το λόγο σε όσους ε, βεβαίως δεν είναι παρόντες εδώ. Και παρόλα αυτά έχουμε αρκετούς ομιλητές και ελπίζω κατόπιν η πατεκπρόσωπος να μπορέσει να πάρει το λόγο. Λοιπόν, πρώτος ομιλητής στη διαδικασία Catch the Eye είναι ο κύριος Αλαφράνκα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μπορεί κανεί να είναι φίλος του Ισραήλ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που ο πρόεδρο των ΗΠΑ κάνει κάτι καινούριο που του έρχεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τρέξει να αλλάξει θέση. Και αυτό ισχύει κυρία Πρόεδρε, για την κατάσταση της Ιερουσαλήμ, την απόφαση 478 του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει να κάνει και με την κυριαρχία στον Κολάν, δηλαδή η απόφαση 2.42 και 4.97 και ισχύει και για την προσάρτηση των ε, επικισμών στη Δυτική Όχθη. Όλα αυτά είναι μονομερή. Το μόνο που κάνουν είναι να διαλύουν τη Διεθνή Συνένεση, να δυσχεραίνουν το διάλογο και την ειρηνευτική διαδικασία που τους ή είναι πολύ περίπλοκη και να καθιστούν ακόμη πιο δυσχερή την επίτευξη της προοπτικής μιας λύσης δύο κρατών που θα συμβιώνουν ειρηνικά σε συνθήκε ασφαλεία που είναι αναγκαίε και για το Ισραήλ και για τον Παλαιστινιακό λαό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Άρνε παρακαλώ. Κυρία Υπατή Εκπρόσωπε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Μογκερίνη και συμφωνώ ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε τα λάθη του Πρόεδρου Τραμπ. Δεν μπορούμε να καταπατάμε το διεθνές δίκαιο να αναγνωρίζεται τον κολάνο Ισραήλ. Με την εκλογή του Νετανιάχου, οι πρόοδοι τη ειρηνευτική διαδικασία δυστυχώ θα σταματήσουν. Διότι αυτό ο Πρωθυπουργό ενισχύει τη σύγκρουση, αναγγέλλοντα ότι θα συνεχίσει την προσάρτηση εδαφών στη Δυτική Όχθη και ότι θα επιβεβαιώσει την ε, προσάρτηση του Γκολάν που ανακοίνωσε πριν τις εκλογές. Οπότε η πολιτική εμπορίου μας έναντι του Ισραήλ πρέπει να εξεταστεί. Η Ευρώπη θα πρέπει εφόσον πρόκειται να είναι μακροπρόθεσμη η πολιτική προσαρτήσεων να αντιπαρατεθεί. Δυστυχώς το Ισραήλ ε, με την πολιτική του και η Αμερική με την πολιτική τους δεν βοηθούν την πολιτική ειρήνευση. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να επιμείνουμε στο διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε. Και επίση δεν θα πρέπει να στείλουμε τους πρέσβεις μας στην Ιερουσαλήμ, όπως έκανε οι Αμερικανοί. Και θα έχει στο πλευρό του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να το κάνει αυτό. Ευχαριστώ κύριε Λίτς. Και τώρα ο κύριος Γκέρικεν. Όλη αυτή η ιστορία με το Ισραήλ έχει να κάνει με το ότι είναι ε, η γη της επαγγελίας ε, το Ισραήλ. Αλλά το Γκολάν και η Δυτική Όχθη μπορούμε να το συζητάμε μόνο αν λάβουμε υπόψη την κατάσταση ασφαλείας του Ισραήλ. Όμως η Ευρώπη ενίσχυσε το Ιράν, το οποίο έχει μπει στη Συρία και ενισχύει τον κίνδυνο που υφίσταται του Ισραήλ στον Κολάν. Η προστασία της Μέκα και της Μεδίνα είναι αυτονόητη. Αλλά όταν πρόκειται για το Ισραήλ, τότε ξαφνικά μιλάμε άλλη γλώσσα. Πρέπει ως Ευρωπαίοι εταίροι να θέλουμε ισορροπία μεταξύ των δυνάμεων και την ειρήνη. Και την ειρήνη όπου γεννήθηκαν οι τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές ε, θρησκείες. Και λόγω της συνολικής κατάστασης έχουμε μόνο έναν αξιόπιστο εταίρο στη Μέση Ανατολή είναι ο εβραϊκό λαός του Ισραήλ. Είναι το μόνο κράτο εκεί που εδώ και χιλιετίε είχε ένα δικαιακό σύστημα που είναι πολύ κοντά στο δικό μας. Και η κατάσταση της ασφαλείας εκεί θα πρέπει να είναι το πρότυπό μας. Δεν έχουν βάση αυτές οι αποφάσεις των ε, ε Ηνωμένων Εθνών. Έχει λήξει ο χρόνος σας λοιπόν. Κύριε Γκέρικ, έχετε ένα, όχι ένα μισή λεπτό. Επόμενος ομιλητής. Η κυρία Ρόζα Νταμάτου, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και σε αυτή την τελευταία ολομέλεια βρισκόμαστε να μιλάμε για την ε, παραβίαση από πλευράς, για την, από την αποδοχή από πλευράς της Αμερικανικής κυβέρνησης, παραβίασης από πλευρά του Ισραήλ, του διεθνούς δικαίου. Έχουμε να κάνουμε με 25.000 δρούζους και 20.000 επίκους από το Ισραήλ σε ένα εδαφός όπως είναι τα υψηπέδα του Γκολάν αμφισβητούμενο μετά την κατάλληλη από το 1967. Είναι μια κατάσταση η οποία μας ανησυχεί. Έτσι λοιπόν μια λύση δύο λαών και δύο κρατών φαίνεται πια να έχει καταστεί μια ουτοπία, μια χήμερα που μόνο ε, κάποιοι ε, φιλόσοφοι μπορούν να συζητούν. Ε, τώρα πια πρέπει να βρούμε μία λύση η οποία θα κάνει σεβαστό το διεθνές ε, δίκαιο και θα κατα κατασυγάζει τις διαφορές που προέκυψαν πριν από το 1967, θα επιτρέψει να ζουν οι άνθρωποι όχι μέσα στην απόγνωση που έχουμε διαπιστώσει με την καταστροφή των σπιτιών των ανθρώπων αυτών, με την παραβίαση κάθε έννοιας ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πρέπει να στηρίξουμε τις χιλιάδες των αδελφών μας στο η Παλαιστίνη, που είναι η μόνη γνήσια δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια των Παλαιστινίων στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είπατε εκπρόσωπε λέει ο Η διαδικασία της ειρήνευσης είναι σε κρίση εδώ και χρόνια. Η λύση δύο κρατών, δύο εθνών, φαίνεται όλο και λιγότερο πιθανό να επιβληθεί. Η κατάσταση στο Ισραήλ έχει αλλάξει ριζικά στο πλαίσιο αυτό και ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο στρατός έχουν ε, Διατηρεί τι δυνάμει του στην περιοχή, βλέπουμε πω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κρατήσει αποστάσει και μπορεί να έχει ένα ρόλο μεν στην περιοχή, αλλά πρέπει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο. Δεν πρέπει επουδενή να επιτρέψουμε αφενό μεν οι Αμερικανοί να υποστηρίζουν το Ισραήλ, αφετέρου δε η Ευρωπαϊκή Ένωση να φαίνεται πω υποστηρίζει την Παλαιστίνη, του Παλαιστινίου. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει δραστήριο ρόλο ω διαμεσολαβητή και όχι ω μέρο τη διαφορά. Ο κύριος Χριστέ, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Το σώμα μας έχει την ευθύνη να έχει μια αντικειμενική προσέγγιση, ισορροπημένη, γιατί επίκειται και η προσλογική εκστρατεία. Πολύ καλό λοιπόν είναι που συζητάμε για τα υψίπεδα του Γκολάν σήμερα. Αλλά μια συζήτηση για τα υψίπεδα του Γκολάν <clears throat> πρέπει να αναφερθεί και στους σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του Ισραήλ στα βόρεια σύνορά του λόγω της παρουσίας Ιρανών στη Συρία και σιητικών πολιτοφυλακών και της τρομοκρατικής οργάνωσης Εσμπολά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχει ισορροπημένη προσέγγιση πρέπει να δείξει ότι δεσμεύεται για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του Ισραήλ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάνω λάθος. Όταν λέω ότι η συζήτηση δεν εξυπηρετεί κανέναν στόχο γιατί η κατάσταση επιτόπου δεν έχει αλλάξει και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ γνωστή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χριστέα. Ο κύριος ε, Σκρίπεκ παρακαλώ. Πρόεδρε, ακούγονται σήμερα πολλές ε, κατηγορίες ε, εις του Ισραήλ Πολλοί είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι αναφέρονται σε συνέπειες μέτρων που μπορεί να πλήξουν και τους πολίτες του Ισραήλ. Και εδώ θα διαφωνήσω. Επιτρέψτε μου να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Το Ισραήλ έχει δικαίωμα άμυνας και ελέγχου και της δυτική Όχθης και των υψηπέδων του Γκολάν που είναι νευραλγικό σημείο μέσα από το οποίο, ε, με βάση το οποίο πολλές εχθρικές στο Ισραήλ δυνάμεις μπορούν να του επιτεθούν. Ξέρουμε από την ιστορία των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χεσμολάχ από την περιοχή αυτή ότι είναι ένας κίνδυνος πραγματικός που δεν μπορεί να αγνοήσει το Ισραήλ. Πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια για το καλό των πολιτών του. Τα νούμερα άλλωστε είναι πολύ εύγλωτα. σε σχέση με τις ε, σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. 200.000 είναι οι Άραβες που απασχολούνται σε Ισραηλινές επιχειρήσεις με πολύ καλούς μισθούς. Ο κ. Παπαδάκης έχει το λόγο. Παπαδάκης. Γνώριση του, της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και την εκεί μεταφορά της Αμερικάνικης πρεσβείας αποτελεί πρόκληση πρώτου μεγέθους η αναγνώριση των κατεχόμενων υψήπεδων του Γκολάν που άρπαξε το Ισραήλ από τη Συρία το 1967 πρόκειται για κινήσει αναβάθμιση των αμερικάνικων συμφερόντων στη μέση ανατολή και στη συρία και στήριξη τη εγκληματική πολιτική του ισραήλ έναντι των ανταγωνιστών του πρωτίστω τη ρωσία για τον έλεγχο των αγορών των πλουτοπαραγωγικών πηγών σε βάρο των λαών τη ευρύτερη περιοχή τεράστιες είναι ευθύνες και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που με την ανοχή των άλλων αστικών κομμάτων στην Ελλάδα εξεπλένει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και προκλητικά απορρίπτει την υλοποίηση της απόφασης της Ελληνικής Βουλής για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους αναβαθμίζοντας όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση τις πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές σχέσεις του Ισραήλ σαν να μην τρέχει τίποτα. Να σταματήσει λοιπόν τώρα η κατοχή του Γκολάν από το Ισραήλ, να δυναμώσει αλληλεγγύη στο Παλαιστινιακό λαό για άμεση η αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την ανατολική ιερουσαλήμ στα σύνορα του 67. Ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη. Τώρα κυρία εκπρόσωπε έχετε το λόγο. Να δηλώσω εκ νέου σαφώς αυτό που έχω ήδη νομίζω δηλώσει επανελειμμένα ε, σε αυτό το ημικύκλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει το Ισραήλ και τους Ισραηλινούς ως εταίρους και φίλους και βλέπει, θεωρεί τους Παλαιστινίους ε, επίσης ως εταίρους και φίλους και τους Αμερικανούς φίλους μας τους βλέπουμε ως εταίρους και φίλους. Αυτό δεν σημαίνει πως οι θέσεις μας, οι πολιτικές μας ε, ε, καθορίζονται αλλού. Ε, καθορίζονται επί τη βάση αυτού που πιστεύουμε ότι είναι προς το συμφέρον της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, που είναι και η δική μας ευρωπαϊκή περιοχή και με το σεβασμό των διεθνών αρχών και δικαίου. Αυτό δεν αλλάζει. Το να επιβεβαιώσουμε εκ νέου και με ενωμένο τρόπο τη θέση μας δεν σημαίνει ότι είμαστε εχθρικοί προς τους συνομιλωτές μας ή τους εταίρους μας που εντωμεταξύ έχουν αλλάξει τη θέση τους. Με, σημαίνει ότι είμαστε επεπισμένοι και έχουμε εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι ανέκαθεν πιστεύαμε ότι η δύναμη του ισχυροτέρου δεν είναι μια καλή αρχή επί της οποίας να βασίζει κανείς την πολιτική του. Η ιδέα ότι μπορείς να αλλάζεις ε, ε, την τάξη με τη χρήση της στρατιωτικής δύναμης είναι επικίνδυνη στην Ευρώπη, στην Ένωση Ανατολή και οπουδήποτε αλλού. Και γι' αυτό και το θέμα, για το θέμα το υψηπέδου του Γκολάν ήμασταν σαφείς. Πιστεύουμε πως οι διεθνείς κανόνες το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς προδιαγραφές πρέπει να τηρηθούν. Και αυτή είναι μια αρχή που είναι προς το συμφέρον όλων. Πολύ συστηματικά και με συνέπεια να στηρίζεται αυτή η αρχή. Αν πιστεύετε